Σας ευχαριστώ. Αρχίζουμε. Πρώτα απ' όλα, καλώς ήρθατε σε αυτή την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. Το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι ε, τα συμπεράσματα από τη συνεδρίαση των συντονιστών. Οι αποφάσεις των συντονιστών σήμερα το πρωί έχουν ως εξής επιβεβαιώνουν τα ονόματα των εισηγητών από την προηγούμενη θητεία και τις υπόλοιπες εκθέσεις από την προηγούμενη θητεία αναθέτονται στους εξή. Η ισορροπία μεταξύ των δύο φίλων σε εκτελεστικές θέσεις, χρηματιστήρια κτλ. Εισηγητής θα είναι η Τζάκι Jones. Ε, πληροφορίες φορολογικές κλπ. Εισηγητής θα είναι ο κ. Γκαρθία Μπλάνκο και νομοθεσία που εφαρμόζεται σε τρίτες πλευρές, cost B. Αυτοί θα είναι οι συγητέ λοιπόν για αυτά τα θέματα. Επίση, οι συντονιστέ αποφάσισαν να μην γνωμοδοτήσουν για υποθέσει που έχουν να κάνουν με την Επιτροπή, εκτό από την απαλλαγή του Γενικού Προπολογισμού του 2018 και θα αποφασιστεί ποιο θα είναι συντάκτη γνωμοδότηση στην επόμενη συνεδρία των συντονιστών. Επίση, οι συντονιστέ ενέκριναν την επιστολή τη διάσκεψη των Προέδρων όσον αφορά για τη σύγκρουση συμφερόντων, όσον αφορά τι επιτροπέ. Η κυρία Κάτρι Σίμψον και η κυρία Πάσκο είναι υπεύθυνοι για αυτό το θέμα. Σύμφωνα με τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να κάνει τέτοια εκτίμηση γιατί δεν υπήρξε ε, χαρτοφυλάκιο για τους δύο υποψήφιους επιτρόπους. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα του χαρτοφυλακίου για να μπορέσει η Επιτροπή μας να κρίνει. Τρίτο θέμα, Ευρωπαϊκή Ένωση και η Υπηρεσία ε, Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Ο Ζωμαρή Καβαντά, που είναι μέλος της 8ης θητείας, θα κληθεί στις 19 Σεπτεμβρίου να έρθει και θα ενημερώσει στις 20 στις 19 Σεπτεμβρίου στη συνεδρίαση της Επιτροπή μας και μετά και τον Οκτώβριο. Συμφώνησαν επίσης οι συντονιστές να προσκαλέσουν τον εκτελεστικό διευθυντή της Υπηρεσίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας στην συνεδρίασή μας στις 14 Οκτωβρίου του 2019 και εγκρίναμε και την ενημέρωση των καθεδρίων γραμμών για τις διαμάχες και αποφάσισαν επίσης να γνωμοδοτήσουμε σε επιστολή που έχει να κάνει με την ε, αναφορά 0660-2018 εκ μέρους ε, Ισπανική επίτροπή για ανήλικέ που βρίσκονται υπό κυδαιμονία. Επίση, συμφώνησαν οι συντονιστέ να προσκαλέσουν εκπροσώπου τη Επιτροπή για να μα παρουσιάσουν τι νέε του προτερότητε όσον αφορά την πνευματική ιδιοκτησία. Και αποφασίσαμε στι 19 Σεπτεμβρίου του 2019 να έχουμε έκτακτη συνεδρίαση και να χρησιμοποιήσουμε τη γραπτή διαδικασία για θέματα που έχουν να κάνουν με τις ακροάσεις των προτινόμενων επιτρόπων. Έτσι συνοψίζονται οι αποφάσεις των συντονιστών. Και τώρα περνάμε στο σημείο 2. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Τώρα θέλω να σας ενημερώσω ότι το πρώτο τμήμα της συνεδρίασής μας είναι και κλεισμένο των θυρών και από το σημείο 5 και μετά θα υπάρχει αναμετάδοση στο διαδίκτυο. Οι χρόνοι που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη είναι καθαρά ενδεικτικοί. Λοιπόν, να διακόψουμε δύο λεπτά τώρα. Όχι, α, όχι ακόμα. Α, άλλο ένα θέμα, το οποίο δεν είναι και κλεισμένο των θυρών ακόμα. Είναι θέματα επικουρικότητας, αλλά δεν υπάρχουν ανακοινώσεις της Προέδρου για αυτά. Και έτσι τώρα περνάμε στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης, που είναι ενέργειες τη Ένωση μετά την προσχώρησή τη στην πράξη τη Γενέβη, τη Συμφωνία τη Λισαβόνα για τι ονομασίες προέλευση και τι γεωγραφικές ενδείξει. Πρόκειται για εξέταση του διορθωτικού. Μετά την έγκριση του Κοινοβουλίου στις 16 Απριλίου του 2019 της θέσης του σε πρώτη ανάγνωση, το κείμενο πέρασε από έλεγχο στους νομικούς γλωσσολόγους προκειμένου να υπάρξει προσαρμογή. Έχουμε το διορθωτικό τώρα που έχει κυκλοφορήσει. Σύμφωνα με, τον, με το άρθρο του κανονισμού 241, η Επιτροπή μας θα εξετάσει το σχέδιο αυτό διορθωτικού και θα αποφασίσει αν είναι ικανοποιημένοι ή όχι προκειμένου να αποσταλεί στην Ολομέλεια. Είμαστε ικανοποιημένοι. Δεν βλέπω να έχει κανείς αντίρρηση, οπότε υποθέτω ότι είμαστε ικανοποιημένοι και θα το στείλω. Α, παρακαλώ κύριε Λεμπρετό. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Διάβασα προσεκτικά το διορθωτικό αυτό το κείμενο απομακρύνεται πολύ από το αρχικό όμω. Δεν πρόκειται απλώς για διορθωτικό. Αν δούμε τις αιτιολογικές σκέψεις υπάρχουν 18 για παράδειγμα, ενώ πριν είχαμε 11. Άρα έχει ξαναγραφτεί το κείμενο και επί της ουσίας επίσης. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές, όπως για παράδειγμα στο άρθρο 6 ε, αναφερόνται τέσσερις μήνες για ενστάσεις αντί για δύο όπως προβλέπονταν πριν. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Εδώ θα μπορούσα να σας αναφέρω πάρα πολλά παραδείγματα. Οπότε με εκπλήσει που έτσι στα γρήγορα εξετάζουμε ένα έγγραφο το οποίο τελικά διαφέρει ουσιοδός από το αρχικό. Για μένα, όταν πρόκειται για διορθωτικό, ε, πρόκειται για μικρές διορθώσεις, ενώ εδώ έχει ξαναγραφτεί από την αρχή με τροποποίησης επί της ουσίας το κείμενο. Αυτό ήθελα να πω. Οπότε εγώ διστάζω, δεν με ικανοποιεί αυτή η διαδικασία. Πιστεύω ότι εδώ δεν παίζουμε το ρόλο για τον οποίο βρισκόμαστε εδώ. Πρόεδρος. Καλώς. Άλλος κανείς ανησυχεί για το κείμενο αυτό. Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι όταν ένα έγγραφο πρέπει να επαναξεταστεί απλά και μόνο για να ε, εξεταστούν οι γλωσσικές δυσκολίες έτσι ώστε να υπάρχει απόλυτη ακρίβεια τουλάχιστον από νομική πλευρά να προταθεί δηλαδή μία ερμηνεία αντί άλλη. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι δυνατόν να συντάξουμε ένα νέο κείμενο γιατί από ό,τι είδα εγώ σε αυτό το νέο κείμενο υπάρχει μία επέκταση, μία διεύρυνση αυτών που είχαν γραφτεί στο αρχικό κείμενο. Και γι' αυτό το λόγο και εγώ δηλώνω ότι είμαι λιγάκι προβληματισμένος όσον αφορά σε αυτή τη νέα ερμηνεία. Και θα ήθελα και οι αρμόδιοι να μου επιβεβαιώσουν ότι πράγματι έχω δίκιο. Ότι δηλαδή όταν πρόκειται για μια ε, νομική διόρθωση καθαρά γλωσσική, στην περίπτωση αυτή ε, δεν μπορούμε να έχουμε μια ευρύτερη ερμηνεία με βάση το αρχικό κείμενο. Ευχαριστώ πολύ. Okay, so we have had two... Ωραία. Δύο έχουν εκφράσει κάποιους δισταγμούς όσον αφορά το κείμενο, γιατί λένε ότι είναι πολύ διαφορετικό από το αρχικό. Οπότε, ή συνεχίζουμε Υποθέτοντα ότι οι υπόλοιποι δεν θεωρούν ότι διαφέρει πολύ το κείμενο ή μπορούμε να το επαναφέρουμε στην επόμενη συνεδρίασή μα για να το επανεξετάσουμε. Λοιπόν, δεν ξέρω, οι άλλοι ευρωβουλευτέ τι έχουν να πούνε. Εγώ θέλω να τονίσω πάντως ότι αυτό που κάνουμε τώρα είναι ότι αποφασίζουμε για να το στείλουμε όχι στην Ολομέλεια. Έτσι καλώς στην Ολομέλεια θα συζητηθεί εκ νέου. Όχι. Α. Παρακαλώ κύριε Βόλκαν. Ευχαριστώ. Εγώ προτείνω να συνεχίσουμε σήμερα. Νομίζω ότι το διορθωτικό σέβεται το πνεύμα της τελικής συμφωνίας στην οποία είχαμε καταλήξει, γι' αυτό και δεν εκφράζουμε εμείς ε, καμιά ανησυχία. Οπότε διαφωνώ με την ε, πρόταση για επανεξέταση. Άλλος κανείς? Ακούσαμε απόψεις και από τις δύο πλευρές, οπότε μάλλον πρέπει να ψηφίσουμε για να αποφασίσουμε αν θα προχωρήσουμε και θα πάει στην Ολομέλεια ή θα το αναβάλουμε και θα το ξανασυζητήσουμε στην επόμενη συνεδρίασή μας. Οπότε θα ψηφίσουμε για την έγκριση του διορθωτικού. Ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε.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 Okay, if there's one question, we will... Λοιπόν, ε, θα ακυρώσουμε την ψηφοφορία, θα ακούσουμε την ερώτηση, γιατί υπάρχει μια ερώτηση από ό,τι φαίνεται. Παρακαλώ, κύριε Λεμπριτού. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η ερώτηση για την οποία ψηφίζουμε. Η ερώτηση είναι να πάει στην Ολομέλεια ή να αναβληθεί. Ψηφίζουμε κατά πόσο εγκρίνουμε το διορθωτικό. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα προωθηθεί στην Ολομέλεια. Οπότε αν θέλετε να πάει το διορθωτικό στην Ολομέλεια ψηφίζετε ναι, υπέρ. Λοιπόν, αρχίζει η ψηφοφορία. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρα τη ψηφοφορίες. Έχουμε το αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα είναι ότι θα προωθηθεί το διορθωτικό στην Ολομέλεια. Ωραία. Τώρα συνεχίζουμε. Τώρα περνάμε σε κεκλεισμένο το θυρών Σε Δύο λεπτά διακοπή προκειμένου να βγουν από την αίθουσα όσοι δεν έχουν δικαίωμα να βρίσκονται μέσα στη συνέχεια.